hey, colleagues, maybe we can make a start if people can take their seats. So apologies for keeping people a little bit delayed because we were having a coordinated meeting. Λοιπόν, καθυστερήσαμε λόγω των συντονιστών. Έχουν αλλάξει πολλά στην Επιτροπή μας και χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο. Ε, τώρα για, το, για την ε, κοινή κοινοβουλευτική, αυτό θα συζητηθεί το απόγευμα. Σήμερα έχουμε ένα θέμα, το πλαίσιο ανάπτυξης, ε, το σφαιρικό, το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015. Θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων πάνω σε αυτό το θέμα και το απόγευμα θα ψηφίσουμε από αυτού και για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Είχαν κατατεθεί 466 τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό φυσικά το θέμα για την Επιτροπή μας, γιατί του χρόνου θα ορίσουμε το νέο πλαίσιο για το αναπτυξιακό για μετά το 2015. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ντάβο Στίερ, τον εισηγητή μας, ο οποίος ήρθε σε εντατικές διαπραγματεύσεις με τους Κιώδης, δούλεψαν όλοι πάρα πολύ σκληρά και κατέληξαν σε ορισμένες συμβιβαστικές λύσεις για το πρόγραμμα του 2015 και η Επιτροπή μας θα μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη άποψη ε, για να παρουσιάσει το Δεκέμβριο στους Υπουργούς την πρότασή της. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Στίερ και μετά στους Σκιώδης και θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντάβο έχει το λόγο πρώτος. Mm. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας και τους Σκιώδης εισηγητές για την καλή δουλειά που έκαναν. Είχαμε αρκετά περίπλοκα πράγματα, 400 66 τροπολογίες. Χτες καταφέραμε να τελειώσουμε και να έχουμε την ακριβή διατύπωση επί της οποίας συμφωνούν οι διάφορες πολιτικές ομάδες για 17 συμβιβαστικά πακέτα. Έτσι διευκολύνεται βεβαίως ο κατάλογος ε, ψηφοφορίας και βεβαίως θα στείλουμε και ένα σαφές μήνυμα. Αυτό το καταφέραμε με έναν τρόπο που ενσωματώνει τις διάφορες απόψεις της Επιτροπής από τις διάφορες πολιτικές ομάδες με έναν πολύ ισορροπημένο τρόπο και βεβαίως απαιτεί απαιτούσε ε, ε, αρκετή καλή θέληση για συμβιβασμούς και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους γι' αυτό. Επίσης ε, σημαντικό για το κείμενο που περιέχεται είναι πως συμπεριλαμβάνουμε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών σε πολλές συμβιβαστικές ε, τροπολογίες και βεβαίως δεν μπορέσαμε να τις δεχτούμε όλες γιατί ήταν άλλες 60 που ήταν σχεδόν τόσο, με, τόσο πολλές ως ε, και η έκθεσή μας. Οπότε τις συμπεριλάβαμε στις συμβιβαστικές αντί για να κάνουμε μια ψηφοφορία μπλοκ. Αλλά σημαντικό είναι και προέκυψε από τις συζητήσεις πως δώσαμε πολύ περισσότερο βάρος ε, και στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Μαζί βεβαίως με τη φτώχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη ως ε, τα βασικά ζητήματα. Βεβαίω επίσης αλλάξαμε κάπως και την δομή της έκθεσης ε, και αντικατοπτρίζει τώρα τις απόψεις των πολιτικών ομάδων ε, για να τονίσουμε ακριβώς με αυτή την παγκόσμια εταιρική σχέση, κάτι το οποίο είχαμε τονίσει σε διάφορα σημεία της έκθεσης, αλλά τώρα θα το τονίζουμε ακόμη περισσότερο. Εδώ πέρα λοιπόν ενσωματώσαμε τα σημαντικά πράγματα για τους συναδέλφους. Συνολικά νομίζω πως τονίζουμε την αρχή της οικουμενικότητας ε, και λέμε πως πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές μας, να λαμβάνουν επίσης υπόψη τους νέους στόχους της βιωσιμότητας και βρήκα μια νέα αποδεκτή λύση ε, στο δίλημα του εάν θα υπάρξει απλοποίηση των στόχων ε, των αναπτυξιακών ή ε, επειδή ίσως εάν ανοίξουμε το πακέτο κάποιοι στόχοι σημαντικοί φύγουν βρήκαμε μια διατύπωση που λέει συμφωνούμε με τη δουλειά της ανοιχτής ομάδας εργασίας ε, αλλά όχι εις βάρος των πιο καινοτόμων στόχων ε, και οπωσδήποτε όχι εις βάρος της προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελευταία παρατήρηση. Τώρα υπάρχει ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο βέβαια εξαρτάται και από τις χτεσινές συμφωνίες ε, ε, μια συμφωνία η οποία νομίζω δεν ε, ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές κάποιας πολιτικής ομάδας, αλλά βεβαίως ε, όλες επέδειξαν καλή θέληση για να πάνε αυτές οι κόκκινες γραμμές όσο δυνατόν πιο μακριά από το κέντρο, για να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερη ουσία στο κείμενο αυτό. Εάν το καταφέρουμε αυτό, το απόγευμα στην ψηφοφορία και είμαι σίγουρος πως θα το καταφέρουμε. Νομίζω πως ε, τώρα ερχόμαστε στην Ολομέλεια με ένα ισορροπημένο κείμενο και με ισχυρά μηνύματα που θα επηρεάσουν την απόφαση του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνατε. Είδαμε τις συμβαστικές προτάσεις με το πρωί με το email. Ωραία, περνάμε στους κοιόδης εισηγητές. Irish Life Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθεια που έκανε. Με 466 τροπολογίες και με πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή του η δουλειά του ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους άλλους κοιόδης με τους οποίους είχαμε μια σωστή συνεργασία στην προσπάθεια της επίτευξης του κοινού στόχου. Μια ισχυρή, εν πάση περιπτώσει, θέση επηρεασμού του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Τα συμπεράσματα του Open Working Group είναι η βάση των συζητήσεων τις οποίες κάναμε και ελπίζω να μπορέσουμε να επηρεάσουμε κάπως τα πράγματα και να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να μην θέσουμε σε κίνδυνο τους πιο φιλόδοξους και καινοτόμους στόχους που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας. Εμείς λοιπόν και το, την καθολικότητα του πλαισίου είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε και τον κατευθυντήριο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της εκρίζωσης της πείνας και της μείωσης των ανισοτήτων ανάμεσα στις χώρες. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά βλέπουμε ότι και οι άλλες πολιτικές ομάδες έκαναν την ίδια επιλογή προτεραιότητας. Νομίζω ακριβώς ε, υπογραμμίσαμε και τη σημασία της επιμονής στα ανθρώπινα δικαιώματα για τους πλέον ασθενείς. Υπογραμμίσαμε τους στόχους στην υγεία, στην εκπαίδευση, ε, στην εκπαίδευση στον τομέα της, του γενετήσιου προσανατολισμού ε, και της ευθύνης των κυβερνήσεων στα πλαίσια της καταπολέμησης της φτώχειας. Είναι μια ισχυρή έκθεση, είναι μια ισόρροπη έκθεση, είναι μια εύθετη χρονικά έκθεση. Και από πλευρά της Επιτροπής Γυναικών υπογραμμίζεται ο κεντρικός ρόλος ο οποίος δίδεται στις γυναίκες και η ουσία της γνωμοδότησής μας περιλαμβάνεται πλέον στην προσπάθεια που κάναμε. Είμαστε για μια ακόμη φορά ικανοποιημένοι. Ελπίζουμε στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή να υποστηριχθεί από τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Και δεν θα μείνουμε εδώ, είναι μια έκθεση την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε προς τους συμπολίτε μας, προς τις κυβερνήσεις μας, πέρα από τους στίχους του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε εμείς στις προτεραιότητές μας μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 όταν τότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Δίβα. Ε, δεν θέλω το λόγο στην παρούσα φάση. Πάβο. και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τάβο και τους υπόλοιπους ε, σκιώδης και την ομάδα της Άλντε και, ε, και για τις τροπολογίες συμβιβαστικές της γραμματείας. Έχουμε ένα πρόβλημα όμως. Η περιβαλλοντική αηφορία. Δεν την έχουμε ασχοληθεί αρκετά με αυτήν. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν έχει εκδώσει γνωμοδότηση η Επιτροπή Ένβη. Αν το έκανε αυτό θα είχαμε πολλές τροπολογίες σχετικά με το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω την στήριξή σας για τρεις τροπολογίες οι οποίες δεν καλύπτονται από τις συμβιβαστικές. Δύο από αυτές ασχολούνται με θέματα της αστικοποίησης 27 και 173. Έχουμε 7,5 δις στον κόσμο και οι μισοί ζουν στις πόλεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθυσμός θα φτάσει περίπου τα 9 δις και τα 2 τρίτα τότε θα ζουν στις πόλεις. Οι μεγαλύτερες πόλεις θα φτάσουν περίπου τα 100 εκατομμύρια κόσμο. Αυτό δεν είναι βιώσιμο οικολογικά και οικονομικά. Γι' αυτό λοιπόν κατέθεσα τις τροπολογίες αυτές πρώτον για να μας υπενθυμίσω το τι μας περιμένει και δεύτερον για να ζητήσω οι περιφερειακές πολιτικές να είναι σε θέση να αντισταθμίσουν την ανάπτυξη αυτή στον κόσμο έτσι ώστε να, να αναπτυχθεί το πρότυπο των μικρότερων αστικών περιοχών και πόλεων. Έχουν προωθηθεί από ορισμένου ε, οι στόχοι της χιλιετίας για τις πόλεις και τις μικρότερες πόλεις. Νομίζω οι τροπολογίες αυτές να γίνουν δεκτές και μία τρίτη τροπολογία Η 165, μπορώ να σας την διαβάσω, είναι σύντομη και ελπίζω να γίνει δεκτή. Ζητάμε την προώθηση της οικολογικής αηφορίας και στις αναπτυγμένες χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι απαιτείται μια τέτοια ισορροπία για να ενισχυθεί η οικολογική διάσταση και αηφόρια. Κατά τα άλλα υποστηρίζουμε όλες τις συμβιβαστικές. Ζητάμε τη στήριξή σας όμως αυτές τις τρεις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Τέβα, να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους της Λόλα Σάντσες ε, ε, από τους ποδέμους από την περιοχή της Καρταχένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Στήρ για τη θαυμάσια έκθεση. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τις περισσότερες τροπολογίες, αλλά υπάρχει πρόβλημα στην παράγραφο 27 για την, το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, είναι υπό τον τίτλο «Πώς θα κινητοποιήσουμε, πώς θα βρούμε κάποιους οικονομικούς πόρους». Έχουμε πρόβλημα πραγματικά εδώ. Δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Καλύτερο θα ήταν να μην υπήρχε αυτό το σημείο στην έκθεση. Μπορώ να ζητήσω από τον εισηγητή να κάνει κάτι. Εκτός αυτού, θαυμάσια η έκθεσή σας. Κύριε Τώρα θα δώσω το λόγο σε άλλους ομιλητές. Πολύ θέλετε το λόγο. Η Λόλα Σάντζος από την ΚΟΕ θα είναι πρώτη γιατί δεν ακούσαμε καθόλου άτομα από την ΚΟΕ. Πριν ξεκινήσεις και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να ζητήσουν το λόγο για να καταγράψουμε Ας γράψουμε τα ονόματα πρώτα και να ξεκινήσει η Λόλα. Ευχαριστώ πολύ. Η Γκουε θα υποστηρίξει το τελικό αποτέλεσμα της έκθεσης αυτής. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε τρεις βασικές ιδέες, τις οποίες εμείς θα θέλαμε να εμείνουμε να συμπεριληφθούν. Η πρώτη είναι ακριβώς ε, η ιδέα του, της καθολικής διάστασης αυτής της προσπάθειας η οποία θα συμπεριλάβει και τις αναπτυγμένες χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες και την καταπολέμηση των ανισοτήτων και ε, των ανισοτήτων λοιπόν σε όλες τις χώρες είναι το κέντρο των, τους, είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να υπάρξει αναφορά στις αιτίες των διακρίσεων και πιστεύουμε ότι ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι το θεμέλιο της προσπάθειας μας. Νομίζω ότι έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ακριβώς και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών που είναι απαραίτητη προϋπόθεση ε, για, την, για τον σεβασμό των δικαιωμάτων γενικά των πολιτών. Είναι πάρα πολύ θετική η ε, πρόταση η εισήγηση της Επιτροπής Γυναικών είναι ένα ιστορικό βήμα και σε σχέση με τα δικαιώματα της, του γενετήσιου, τα αναπαραγωγικά. Νομίζω ότι εφόσον γίνει δεκτή η πρόταση αυτή θα είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Στήρ, να ευχαριστήσω και την ομάδα του. Εμείς εμένουμε πάντως αυτές τις τρεις προτεραιότητες ε, λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια ευρύτερη γενικότερα ε, συμφωνία η οποία θα ενίσχυε γενικότερα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Άλλοι τέσσερις θέλουν το λόγο, θα διαβάσω τα ονόματά τους και αν κάποιος θέλει το λόγο να το πει τώρα. Σαλόμ, σοσιαλιστές, μάλλον Μπεσερίλ από το ΕΛΚ, Σαλόμ, Αλιό, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ενδιάμεσα θέλει το λόγο. Χιμένες Μπεσερίλ. Ε, Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω και εισηγητά για τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε για να ολοκληρώσετε σε τόσο σύντομο χρόνο μια τόσο πλήρη έκθεση και με τόσο υψηλό αριθμό τροπολογιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το συνενετικό πνεύμα σας που οδήγησε σε μια πραγματικά ισορροπημένη λύση. Να ευχαριστήσω και όλους τους κοιόδης εισηγητές, οι οποίοι ε, πήρα και εγώ μέρος ε, για το θέμα της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γυναικών. Σας ευχαριστώ για τη συμπερίληψη της ε, γνωμοδότησης αυτής, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά θετικά και στον τομέα τον κοινωνικό και στον τομέα των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για μετά το 2015. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε πλήρως διευκρινιστεί από πριν. Επίσης είναι θετικό το συμπεριλάβαμε την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών, των παιδιών, του γενετήσιου ακροτηριασμού, των υποχρεωτικών γάμων. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία υπογραμμίζει η σημασία η ίδια της ύπαρξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Και τέλος, έχει μεγάλη σημασία και άλλο ένα θέμα για τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε εμείς όλα αυτά τα θέματα και ιδιαίτερα το θέμα της καταπολέμησης της φτώχειας αν δεν εμπλέξουμε και τις τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστώ και ε, συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά. Σαλόμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Στήρ για μια τεράστια προσπάθεια. Εγώ συμμερίζομαι πολύ στις θέσεις τις οποίες ε, εξέφρασε η συγγήτρια της πολιτικής μας ομάδας. Όχι ότι συμφωνούν κανείς πάντα με αυτά τα οποία λέει ο εισηγητής της ομάδας του, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό συμβαίνει. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Στήρ για την αποδοχή τριών αλλαγών, αν θέλετε, τριών ε, υποθεμάτων τα οποία ε, έχουν συμπεριληφθεί. Και όχι μόνο γιατί εγώ επιμένω σε αυτά, αλλά γιατί πιστεύω ότι είναι τομεί στους οποίους μπορούμε να έχουμε ε, μια ενισχυμένη πολιτική παρέμβαση. Ένας από τους τομείς αυτούς είναι το θέμα των ανθρώπων με κάποιες μορφές αναπηρίας θα πρέπει στα πλαίσια των στόχων εμείς με εγκάρσιο τρόπο να θεωρήσουμε το θέμα αυτών των ανθρώπων που είναι ένα σοβαρό ποσοστό σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπου δεν υπάρχουν προληπτικές πολιτικές και υπάρχει ψηλότερος κίνδυνος αναπηρίας. Δεύτερον, Το θέμα της ανθρωπιστικής απάντησης είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί ε, στους στόχους σας. Και τρίτον, να συνδέσουμε την στήριξη της οικονομικής διακυβέρνησης ε, σε σχέση με τις χώρες οι οποίες έχουν ε, αποτύχει οργανωτικά και τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται μετά το τέλος των σειράξεων. Οι χώρες αυτές αναδύονται με πάρα πολύ ε, εύθραστη την κατάσταση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Τώρα για την αναπαραγωγική υγιεινή και υγεία. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πάλι ότι, ε, και αυτό ακούστηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους, ότι χρειάζεται να δοθεί ένας αγώνας, ο αγώνας αυτός θα πρέπει να είναι συνεχής, εμείς έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες, εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να είμαστε αδρανείς, εμείς επιμένουμε στα πλαίσια των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών και η συζήτηση αυτή είναι μια ευκαιρία για να πούμε ότι εμείς επανειλημμένα και στις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδου υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτά των γυναικών. Είχαμε κάνει και την έκθεση για τις, ε, το 2010 για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες και θυμάμαι ότι είχε περάσει με πάρα πολύ μικρή διαφορά, 290 περίπου ψήφοι ε, υπέρ και 260 τόσες κατά. Εμείς ε, πολλές φορές έχουμε διαφορετικές απόψεις, διστάμενες απόψεις, αλλά καταφέρνουμε να υποστηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Δεν είχα το όνομά σας ότι ήσασταν σκιώδης εισηγήτρια, έχετε το λόγο τώρα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά είχε φτάσει η στιγμή για αυτή την έκθεση. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι παίρνω το βάπτισμα του πυρός ως κοιόδηση εισηγήτρια. Νομίζω καταβάλαμε κάθε προσπάθεια και έτσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τόσο σύντομα μια τόσο μεγάλη έκθεση. Νομίζω πως ε, πραγματικά βασιστήκαμε στο, σε αυτά τα οποία έλεγε η ανοιχτή ομάδα εργασίας του ΟΗΕ, τα οποία αντιγράψαμε στην έκθεσή μας. Αναφέρθηκαν ήδη τα δικαιώματα των γυναικών, ο σημαντικός ρόλος των γυναικών στην αναπτυξιακή συνεργασία και αυτό αναφέρεται εδώ και τα δικαιώματα των παιδιών. Ε, ειδικά βεβαίως ε, τα κορίτσια, οι ευριανές γυναίκες ε, που διαφυλάσσουν τη σταθερότητα σε πολλές περιοχές. Και αυτά τα αναφέρουμε στην έκθεσή μας ανισότητα, υγεία, όλα τα είπαμε. Επίσης αναγνωρίζουμε πως η κλιματική αλλαγή είναι ένας τομέας ε, που θα καθορίσει το μέλλον ε, και τα μελλοντικά προβλήματα και θα πρέπει να τα δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα διασφαλίσουμε την διατροφή Δεν έχει νόημα να το σκεφτόμαστε μόνο όταν γίνεται μια καταστροφή, αλλά να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη διατροφική ασφάλεια σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Και να πω εδώ πέρα τη χωριστή ψηφοφορία που ζητήσαμε εμείς οι πράσινοι, η τροπολογία υπαριθμών 84, γιατί είναι κάτι το γενικότερο, μια γενικότερη πρόκληση. Το περιβάλλον που είναι η βάση της ζωής ε, πρέπει να μας απασχολεί στο μέλλον. Αυτή είναι η διάσταση που χρειαζόμαστε και για τη διατροφή του ανθρώπου. Να τονίσουμε λοιπόν την πτυχή του περιβάλλοντος. Συνολικά συμφωνούμε με την έκθεση αυτή. Είναι μια καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση και πραγματικά είναι κάτι που χρειαζόταν και ευχαριστώ τους συναδέλφους και κυρίως τον κύριο Στίερ. Ευχαριστώ. Θα δούμε την τροπολογία 84. Δεν έχω τον κατάλογο ψηφοφορίας εδώ, δεν ξέρω αν είναι χωριστή ε, ψηφοφορία, θα μου πει η γραμματεία. Είναι χωριστή ψηφοφορία ήδη ωραία, ναι. Ο κύριος Αλλιώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είμαστε στις 11 Νοεμβρίου. Ε, θέλω να τιμήσουμε όλους αυτούς που έπεσαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην έκθεση υπάρχουν δύο καλά πράγματα, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα που λείπουν, που θα μπορούσαν να υπάρχουν και στην αιτιολογική σκέψη. Το πρώτο που είναι σημαντικό είναι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ε, είτε στις σχέσεις βορρά-νότου, είτε ε, από τις χώρες της φτωχές. Ε, μην το ξεχνάμε, γιατί η διαχείρισή τους είναι τμήμα της υφόρου ανάπτυξης. Ένα άλλο θέμα που λείπει και που με εκπλήσει ακόμα περισσότερο, μια και πρόκειται για μια και ο ε, εισηγητή είναι από μια χώρα που συνεισέφερε πολύ σε αυτό το θέμα ε, και δεν λέει τίποτα όμως, είναι η διαφθορά. Ε, πολλά από τα στοιχεία ανάπτυξης που δεν έγιναν, πολλά από την ανάπτυξη που δεν πραγματοποιήθηκε, οφείλεται ακριβώς στη διαφθορά που υπάρχει σε αυτές τις χώρες. Δεν ξέρω αν έχει σταματήσει αυτή η μάστιγα. Θα ήθελα να υπάρχει μια ειδική παράγραφος, όχι μόνο για την ε, παλιά διαφθορά και σημερινή ήδη με τους Αφρικανούς ΕΤΕΡ αλλά και για να δημιουργηθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε τα ίδια στο μέλλον και να ελέγξουμε πού πηγαίνουν τα, τα, τα κονδύλια αναπτυξιακής βοήθειας ε, της Ευρώπης ε, προς χώρες που βρίσκονται σήμερα σε μεγάλη αστάθεια. Δεν βλέπω άλλους συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, εν αυτή περιπτώσει. Α, ο Νάτα. Δεν σας είδα, πάρτε το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτά που μόλις άκουσα είναι αποφασιστική σημασίας. Η διαφθορά είναι ένα από τα βασικά εμπόδια της ανάπτυξης. Οποιαδήποτε βοήθεια που δίδεται σε μία χώρα όπου υπάρχει διαφθορά είναι σαν να βάζεις νερό ας πούμε ε, σε μια τρύπα. Χάνεται. Θα πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη για το ότι θα πρέπει να ελέγχουμε τα αναπτυξιακά κονδύλια και από τη χώρα που ξεκινούν και στη χώρα που φτάνουν. Ε, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι οι πιο διεφθαρμένες. Ε, συχνά αυτές οι χώρες είναι πιο υπανάπτυκτες. Κατά συνέπεια, το να βοηθού, βοηθάμε τις πιο υπανάπτυκτες ε, χώρες που είναι ταυτόχρονα και πιο διεθαρμένες είναι απλώς ότι εμείς καθησυχάζουμε τις συνειδήσεις μας και ξέρουμε ότι αυτή η βοήθεια ανάπτυξης είναι εντελώς άκυρη, ακυρώνεται. Είναι σαν να μην τη δίνουμε. Στην ε, Γουινέα του Ισημερινού έχει ε, Κατά κεφαλήν, εισόδημα ίδιο με της Πορτογαλίας ή της Ελλάδας. Στην πραγματικότητα βοηθάμε τους κλέφτες εκεί της Γουινέας. Ε, υπάρχουν σε πολλές χώρες αντίστοιχες, ε, αντίστοιχοι κλέφτες στην Αφρική, στο Κονγκό. Τι νόημα έχει η αναπτυξιακή υπαρχουν σε πολλες χωρες αντιστοιχες αντιστοιχοι κλεφτες στην αφρικη στο Κονγκό, σε μια χώρα όπου η διαφθορά την καθορίζει, την προσδιορίζει. Η Νιγερία. Μπορώ να σα δώσω πάρα πολλά ονόματα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, τι ξέρουμε. Ξέρουμε και ποιε είναι οι δείκτε διαφθορά, ας πούμε, αν τον κόσμο. Και εκεί βλέπουμε χώρες οι οποίες ζητάνε βοήθεια. Όμως, θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό για να παρακολουθούμε το που πηγαίνουν τα αναπτυξιακά κονδύλια. Δύο, θα πρέπει να λέμε ότι η, διαφθορά είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της υπανάπτυξης. Και οποιαδήποτε βοήθεια θα πρέπει να ελέγχεται απόλυτα, ούτω ώστε να μην καταλήγει ε, ως συνήθως σε ένα λογαριασμό όψεως στην Ελβετία. Σε ένα τρεχόμενο λογαριασμό στην Ελβετία. Ο κύριος Πρέντα. Όχι, η Κομισιόν. καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση, όχι μόνο λόγω της ουσίας της, αλλά και λόγω της χρονικής στιγμής που υποβάλλεται. Γιατί μας βοηθά να προχωρήσουμε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, τόσο ώστε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα του Συμβουλίου στο επόμενο ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο. Και επομένως η εισφορά του Κοινοβουλίου για αυτή την ιστορία, για αυτή τη συζήτηση είναι σημαντική. Ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις ε, επιταχύνονται στη Νέα Υόρκη και για αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε σύντομα μια ισχυρή ενιαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαπραγματεύσεις. Αυτή η θέση δεν περιορίζεται φυσικά στην, ε, στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και στη μελλοντική ατζέντα, αλλά θα πρέπει να έχει μια στέρεη προσφορά ε, εμείς για τη χρηματοδότηση Ε, στην διάσκεψη της Αντίς που θα γίνει τον επόμενο Ιούλιο. Εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας αρχές του χρόνου, του επόμενου χρόνου. Συζητήσαμε και διάφορα θέματα στις ε, τροπολογίες. Περιμένουμε την πρώτη σύνταξη της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα και δεν ξέρω αν ο Γενικός Γραμματέας θα κάνει προτάσεις για το clustering. Θα δούμε αυτές τις προτάσεις, ελπίζω, πολύ σύντομα. Ο κύριος Στίερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές και όλους όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και μίλησαν για να ακουστούν αυτές οι απόψεις, για να ανταλλαγούν αυτές οι απόψεις. Δύο θέματα έχουν να ακουστεί, με ιδιαίτερη έμφαση. Το πρώτο, η ανάγκη καταπολέμησης διαφθοράς. Εμπεριέχεται απόλυτα στην έκθεση το θέμα αυτό. Φυσικά είχε διάφορες πτυχές η έκθεση αυτή και οι συνάδελφοι μόνο το, κοιτάξαν μόνο το πρώτο σχέδιο της έκθεσης που, ήταν, που περιοριζόταν και από τον αριθμό των λέξεων. Αλλά μέσω των συμβιβασμών και μέσω των τροπολογιών και των συμβασμών σε δύο τουλάχιστον παραγράφους χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη διατύπωση για την ανάγκη καταπολέμησης διαφθοράς και ο τίτλος ε, για μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, μιλάει για τη διαφθορά αλλά και για την καλή διακυβέρνηση ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του προβλήματος. Ή κάποιες από τις ρίζες του προβλήματος που βλέπουμε στην αναπτυξιακή ατζέντα. Φυσικά, για τις χώρες, επιμέρους χώρες, εμείς δεν κατονομάζουμε χώρες στην έκθεση. Ξέρω ότι η Γουινέα του Ισμερινού ε, δεν έχει λάβει οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετό καιρό. Σας διαβεβαιώ όμως κύριοι Ευρωβουλευτές ότι έχουμε ξεκαθαρίσει τις απόψεις μας και μιλάμε για την ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης, στα πακέτα συμβιβασμών δεν μπόρεσαν όλες οι πολιτικές ομάδες να πούν ότι συμφωνούν να τα προσυπογράψουν. Ευχαριστώ την ECR για την ευελιξία της όμως να υποστηρίξει τελικά την έκθεση ως έχει. Νομίζω τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ε, προστατεύονται και αναφέρονται στην έκθεση. Επίσης υπάρχει και ένας κοινωνικός ρόλος της ιδιοκτησίας Εδώ στο Βέλγιο, στο νέο συνασπισμό, γίνεται μια συζήτηση μεταξύ χριστα... χριστιανοδημοκρατών για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πέραν αυτού όμως, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε επί του συνόλου της έκθεσης και σε ευχαριστώ για την ευελιξία σας. Εν τέλει, νομίζω ότι καταλήξαμε σε μία ισορροπημένη έκθεση που συμπεριλαμβάνει τις απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων. Ήμασταν ε, πολύ προσεκτικοί σε ευαίσθητα θέματα. Δεν θέλησαμε να αγνοήσουμε κάποιες κόκκινες γραμμές και να τις περάσουμε, αλλά παράλληλα θελήσαμε να στείλουμε και ένα ισχυρό μήνυμα. Περιμένω λοιπόν την ε, ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ ξανά όλους τους συναδέλφους, καθώς και τη γραμματεία. Και εγώ σε ευχαριστώ κύριε Στυρ για τη δουλειά σας. Θα ψηφίσουμε στις 3 το απόγευμα την έκθεση αυτή. Να υπενθυμίσω ότι το στοιχείο για το JPA το, το βάζουμε μετά τις ψηφοφορίες. Έχουμε χρόνο να ετοιμάσουμε και τους καταλόγους των ψηφοφοριών. Θα τα πούμε στις 3 για τις ψηφοφορίες. Και το σημείο 10 δεν θα το συζητήσουμε τώρα.